συνεδρίαση. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση για το κράτο δικαίου στη Μάλτα, έχω να σα κάνω κάποιε ανακοινώσει. Ε, Καταρχά, όσον αφορά τα πρακτικά τη χθεσινή ε, συνεδρίαση, εγκρίθηκαν, είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν παρατηρήσει. Αν όχι, εγκρίνονται λοιπόν.